Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον άλλο εισηγητή μας, τον κύριο Βλάσακ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και ε, την επικοδομητική συζήτηση. Για να ολοκληρώσω τη συζήτηση θέλω να κάνω δύο προκλητικά σχόλια. Τα διαρθρωτικά ταμεία δημιουργήθηκαν για να εξισορροπήσουμε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Γι' αυτό άλλωστε θα πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους της ε, σύγκλησης και το στόχο 1. Θα ε, υπάρξουν ε, ανάγκες και οποιασδήποτε ε, απόπειρες να δημιουργηθούν κατηγορίες ενδιάμεσες ή να ενισχυθεί ο στόχος 2 θα πρέπει να αποσοβηθούν. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να πάρουμε κονδύλια από τους πλουσίους για να τα ξαναδώσουμε στους πλουσίους με αυτούς τους στόχους. Οι στόχοι ε, είναι διακριτοί ο στόχος 1 και ο στόχος 2. Ε, επίσης πιστεύω ότι είναι κρίσιμο να Ε, σταματήσουμε να πηγαίνουμε κόντρα στην αγορά. Δεν μπορούμε ε, να ε, κάνουμε διακρίσεις εις βάρος κάποιων ενισχύοντας συγκεκριμένους μόνο και εκείνοι που δεν παίρνουν βοήθεια από την Ένωση είναι σε μειονεκτική θέση και μη ανταγωνιστική. Οι τελικοί αποδέκτες θα πρέπει να είναι περιφέρειες, δήμοι, κοινότητες κτλ. οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που να επενδύουν στη συνέχεια σε ε, μέτρα αναπτυξιακά και προγράμματα. Αυτή την κατεύθυνση νομίζω πρέπει να ακολουθήσουμε. Όπως είπε και ο Νίλ Άμστρονγκ, θα είναι ένα μικρό βήμα για τα ευρωπαϊκά ταμεία, αλλά είναι τεράστιο άλμα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η κυρία Σάντσε Σμιτ. Η κυρία Σάντσε Σμιτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα η Ευρώπη είναι σε κρίση. Δημοσιονομική, μακροοικονομική, χρηματοπιστωτική, κοινωνική αλλά και ηθική οι πολίτες βλέπουν στην Ευρώπη ένα εχθρό ε, που ε, τους επιβάλλει δραστική λιτότητα. Δεν κοιτάνε τι κάνει για τις επενδύσεις, για την ενίσχυση της απασχόλησης, για την ένταξη των λιγότερο ευνοημένων και για την κάλυψη των ανισορροπιών και των ελλημάτων μεταξύ των περιφερειών. Θα ψηφίσουμε αργότερα το πακέτο για τη μακροοικονομική διακυβέρνηση που προβλέπει υπεύθυνα μέτρα για την εξυγίαση των δημοσιονομικών, για την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας. Η πολιτική συνοχή είναι ο δεύτερο πυλώνα όπου καλείται να βασιστεί αυτή η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που να συμπεριλαμβάνει, που να είναι ευφυή και βιώσιμη. Είναι ε, οι δύο του ίδιου νομίσματος. Και θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ε, αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε και την πολιτική αυτή και τον προπολογισμό τη και να πείσουμε τα κράτη ότι η περιφερειακή πολιτική δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Τα διακυβεύματα της δημοσιονομικής ε, διαπραγμάτευση για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι πολλά θα πρέπει να είναι η πολιτική μας καλύτερη, πιο απλή, πιο ορατή, με ενίσχυση της εδαφικής ε, συνεργασίας και να απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες. Γι' αυτό ε, υποστηρίζω την πρόταση Πίπερ που ε, είναι να δημιουργηθεί μια ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα στο 75% και 90% του ΑΕΠ της κοινότητας. Έτσι θα μπορέσουν πολλές περιφέρειες που αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα ανάπτυξης να έχουν ίση και ισορροπή μεταχείριση ενίσχυση. Βεβαίως θα ήθελα να επιμείνω και πάλι στη σημασία της ενίσχυσης της ε, δαφικής συνεργασίας στην Ευρώπη, μεταξύ περιφερειών δηλαδή. Είναι η μεταφορά στην πράξη των όσων είπε ο Ρομπέρ Σουμάν, ότι δεν θα γίνει η Ευρώπη διαμιάς, αλλά με συγκεκριμένα βήματα, με ε, μία εκ των πραγμάτων αλληλεγγύη. Αυτά τα είπε πριν από 60 χρόνια και είναι ακόμα τόσο επίκαιρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ε, Τώρα το λόγο έχει ο τελευταίο συγητή μα, κ. Σταυρακάκη. Κύριε αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ όλου του συγητέ των εκθέσεων με τι οποίε μα δόθηκε σήμερα ευκαιρία να συζητήσουμε βασικέ διαστάσει τη μελλοντική πολιτική συνοχή και να εκφράσουμε τι κύριε θέσει μα από αυτόν. Θα ήθελα ωστόσο να σταθώ στην έκθεση του κυρίου Πίπερ, στην οποία ήμουν σκιώδη συγητή, γιατί σε αυτή διατυπώνονται οι αναλυτικέ θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αρχιτεκτονική που θα πρέπει να έχει η πολιτική συνοχή μετά το 2013 να υπογραμμίσω ότι οι κύριε θέσει μα έχουν ήδη διατυπωθεί και εγκριθεί από την ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σε ειδικό κεφάλαιο του ψηφίσματο για τι μελλοντικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ ευρωπαϊκή ένωση που αφορά την πολιτική συνοχή δεν θα κάναμε υποχωρήσει στι θέσει μα αυτέ. η μελλοντική πολιτική συνοχή πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο προπολογισμό προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στι νέε προκλήσει να στηρίζει όλε τι περιφέρειες τη ευρωπαϊκή ένωση με ιδιαίτερη πάντα έμφαση στι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τι περισσότερε αναπτυξιακέ δυσκολίε να περιέχει θεματικούς στόχους αλλά παράλληλα και ένα βαθμό ευελιξίας να στηρίζεται σε απλοποιημένους και όσο το δυνατόν ενοποιημένους κανόνες μεταξύ των ταμείων της και να διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες της ένωσης θα μπορούν να απολαμβάνουν το ωφέλη της ακόμα και αν ζουν στο πιο απομακρυσμένο μέρος της ευρωπαϊκής ένωσης σε νησιά και ορεινές περιοχές τέλο ειδικότερα για την πρόταση τη δημιουργία μια ενδιάμεση κατηγορία στήριξη την οποία τόσο εγώ και η πολιτική μου ομάδα όσο και μια μεγάλη πλειοψηφία του κοινοβουλίου υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνώ απόλυτα με την άποψη που έχει εκφράσει σήμερα ο επίτροπο χαν. η δημιουργία τη είναι απόλυτα δικαιολογημένη και θέλουμε το μελλοντικό σύστημα στήριξη των περιφερειών να αντιμετωπίζει κατά δίκαιο απλοποιημένο και διαφανή τρόπο περιφέρειε που παρουσιάζουν ίδιο επίπεδο ανάπτυξη πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ξεκάθαρο μήνυμα πως η ευρωπαϊκή ένωση ό,τι βλέπουμε πίσω από τα στατιστικά στοιχεία ιδιαίτερα στη συγκυρία της σημερινής οικονομικής κρίσης. ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνεται εδώ η κοινή συζήτηση. Η ψηφοφορία για αυτό το θέμα και για πολλά άλλα ακολουθεί στις 12. Μικρή διακοπή για 12-13 το πολύ λεπτά. Ευχαριστώ. Not with a, not with a cock, I think. No. yes.